if you help me. Okay. Thanks. Good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας παρακαλώ να καθίσετε στις θέσεις σας. It is a privilege to... Είναι ιδιαίτερα Ευχαριστώ για μένα που μπορώ να σας καλωσορίζω. Άρχη της συνεδρίαση. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο στόχος της σημερινής συνεδρίασης είναι η εκλογή του Προέδρου και των Προέδρων βάσει του ε, ανάλογου άρθρου του Καρσό. Σύμφωνα με το άρθρο 87 έχουν ανακοινωθεί οι υποψηφιότητες. Σημειώνω ότι έχουμε απαρτία. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποιον ε, προτείνετε για το Προεδρία της Επιτροπής αυτής. Θα ήθελα να δώσω στον κύριο Ζόντεργκάτ, συντονιστή της ΓΚΟΕ, το λόγο. Ε, ε, Ευχαριστώ. Εγώ εδώ είμαι ε, αναπληρωτής. Θα ήθελα να προτείνω όμως τον κύριο Γκούσταυσον, υποψήφι για την Προεδρία. Ευχαριστώ. Άλλη υποψηφιότητα. Δεν βλέπω να υπάρχει άλλη υποψηφιότητα εδώ. Ο κύριος να από ό,τι κατάλαβα, δέχεται την υποψηφιότητα αυτή. Συμφωνείτε. Thank you very much. I have been... Σας ευχαριστώ πολύ. I declare, I declare Mr. to be... Λοιπόν, ο κύριος Γκούσταυσον είναι ο προνόεος πρόεδρος μας. Σας ευχαριστώ για το μέχρι τούδο έργο σας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Καλή δουλειά τα επόμενα δύο μισή χρόνια. Σας παραδίδω το θόκο του πρόεδρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περάσω στα σουηδικά αν μου επιτρέπετε και αν δεν καταλαβαίνετε χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σας. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε. Πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ καλά που μου δώσατε την εμπιστοσύνη σας όλοι μετά από τουρισμίνες μήνες που είμαι εδώ και ε, σας υπόσχομαι ότι θα εργαστώ σκληρά για την ισότητα των φίλων ούτως ώστε τα θέματα της ισότητας να είναι πάντα επίκαιρα στο Κοινοβούλιο και σε όλες τις αποφάσεις που παίρνουμε να λαμβάνετε πάντα υπόψη η ισότητα. Με τη βοήθεια της γραμματείας και με δική σας συνεργασία, οπωσδήποτε θα συνεχίσω την στενή συνεργασία με όλους. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε. Τώρα θα περάσουμε στην εκλογή των αντιπρόεδρων. Έχουμε απαρτία από ό,τι βλέπω. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία και παρακαλώ να ακούσω τις... ποιος είναι υποψηφίος για την πρώτη αντιπροεδρία. Κύριε Ανέτεζεφ. Ευχαριστώ Πρόεδρο. Θα ήθελα καταρχήν να σας ε, συγχαρώ για την εκλογή σας. Εξ ονόματος του ΕΛΚ ε, θα ήθελα να υποβάλω την υποψηφιότητα της κυρίας Λίβια Ρόκα για την πρώτη αντιπροεδρία της Επιτροπής Γυναικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλο που θα ήθελε το λόγο επ' αυτού, όχι. Έχουμε μία υποψηφιότητα λοιπόν. Η κυρία Λιαγορακά. Μπορούμε διαβοήσει ίσως να την εκλέξουμε. Φαίνεται ότι υπάρχει συνένεση. Θέλει κανένα το λόγο. θα ήθελα να σας πω ότι έχει εκτελέσει το έργο της, έχει υποβάλει δηλαδή τα στοιχεία για τα οικονομικά της συμφέροντα. Με συγχωρείτε, μπερδεύομαι αγγλικά, σουηδικά ανακατεμένα, θα προσπαθήσω να μιλώ μόνο σουηδικά. Είναι πιο εύκολο να επικοινωνήσουμε αν μιλάτε αγγλικά, μου φαίνεται. Θα ακούσω κάποιον που έχει περισσότερη εμπειρία λοιπόν. Η κυρία Γιαρόκα έλεγα έχει συμπληρώσει αυτή τη δήλωση των οικονομικών συμφερόντων, μπορεί λοιπόν να εκλεγεί. Έχουμε ε, μία μόνο υποψήφιο. Διαβοής λοιπόν. Μπορείτε παρακαλώ να περάσετε εδώ, στο βήμα. It's not so easy to take it in English because you don't... Δεν είναι πολύ εύκολο να τα πει κανένα στα αγγλικά γιατί δεν ξέρω τις διαδικαστικές ε, εκφράσεις που χρειάζονται. Βέβαια πιο εύκολο θα μου ήταν σας εδώ, αλλά θα προσπαθήσω, θα προσπαθήσω αφού μου το είπατε. Περνάμε τώρα στην εκλογή του δευτέρου αντιπρόεδρου. Και εδώ έχουμε πάλι ακόμα απαρτία. Οι υποψηφιώτε για τη δεύτερη αντιπροεδρία, παρακαλώ. Το λόγο έχει η κυρία Στρέλα. Α, η κυρία Τόμψον, συγγνώμη. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Για τη δεύτερη αντιπροεδρία θα ήθελα να προτείνω την κυρία Εντίτε Στρέλα. Άλλες υποψηφιότητες υπάρχουν, όχι. Μπορούμε λοιπόν να... Ε, συγγνώμη. Σας ρωτώ κυρία Στρέλα, δεχόσαστε την υποψηφιότητα αυτή. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και σας, και σας ενημερώνω ότι έχει συμπληρώσει την δήλωση για τα οικονομικά της συμφέροντα κυρία Στρέλα. Μπορούμε να πράσουμε στην εκλογή λοιπόν. Μία υποψήφια έχουμε. Μπορούμε διαβοής λοιπόν να την εκλέξουμε. Please take Παρακαλώ, ελάτε εδώ πάνω στο βήμα. Θα περάσουμε λοιπόν στην εκλογή της τρίτης αντιπρόεδρου, του τρίτου αντιπρόεδρου. Και εδώ έχουμε απαρτία, όπως χρειάζεται. Υποψηφιότητες παρακαλώ για την τρίτη αντιπροεδρία της Επιτροπής μας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ελισσοβέ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να προτείνω την κυρία Ελίζα nominations? Άλλες υποψηφιότητες παρακαλώ. Όχι. Να ρωτήσουμε την κυρία Μπορσέτα εάν συμφωνεί να είναι υποψήφια. Μάλιστα, πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Και να σας υποθέσω ότι η κυρία Μπορσέτα έχει ε, σωστά συμπληρώσει την δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Μια που δεν έχουμε άλλους υποψήφιους, μπορούμε νομίζω να εκλέξουμε διαβοήστη Ωραία, περνάμε τώρα στην εκλογή τετάρτου αντιπρόεδρου. Έχουμε την απαραίτητη απαρτία και θα ήθελα να μου υποβάλλετε τι υποψηφιότητε για την τέταρτη αντιπροεδρία τη Επιτροπή μα. Η κυρία Νελέτσεβα έχει το λόγο. Μάλιστα, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να προτείνω την κυρία Μπάρμπαρα Ματέρα. Ευχαριστώ πολύ. Δεχόσαστε την υποψηφιότητά σα. Μάλιστα, Πρόεδρε. Άλλες υποψηφιότητες. Όχι. Ωραία, θα, να σας ενημερώσω ότι και η κυρία Ματέρα έχει συμπληρώσει την δήλωση οικονομικών συμφερόντων και μια που δεν έχουμε άλλους υποψηφίους θα μπορούσαμε νομίζω να εκλέξουμε διαβοή στην κυρία Ματέρα. Thank you very much everybody and... Λοιπόν, σα ευχαριστώ όλου και περνάμε τώρα στην έγκριση τη ημερησία διάταξη. Και τώρα θα μιλήσω σουηδικά. Okay, we have um, uh, Λοιπόν, υπάρχουν παρατηρήσεις για την ημερησία διάταξη. Κύριε θα ήθελα να αλλάξουμε λίγο τη σειρά των ψηφοφοριών. Η πρώτη ψηφοφορία θα είναι οι γυναίκες διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων. Αυτό θα είναι το πρώτο σημείο της ψηφοφορίας. Η κυρία Σοφίντφελτ δεν είναι ακόμα εδώ, οπότε θα πρέπει να αλλάξουμε και τη σειρά των θεμάτων που θα συζητήσουμε. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε τώρα το σημείο 7. Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν παρατηρήσει, εγκρίνει τη ημερησία διάταξη. Τώρα, ανακοινώσει του Προέδρου. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι η κυρία Φιγκερέτο από την ΚΟΕ έχει φύγει από το κοινοβούλιο και την αντικαστά η κυρία Σούπερ που δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι παρούσα σήμερα γιατί εξελέγει αντιπρόεδρος σε μια άλλη επιτροπή. Θα ήθελα να τη χαιρετήσω, αλλά και την κυρία Κοχμερίν θα ήθελα να χαιρετήσω στην επιτροπή μας. Αυτές είναι οι αλλαγές που έχουμε. αυτή τη στιγμή στη σύνθεση της Επιτροπής μας. Κατόπιν, όπως ξέρετε πολλοί από εσά, η Σαμπίνα δεν θα συνεχίσει να συνεργάζεται εδώ μαζί μας, γιατί από το 1 Φεβρουαρίου και μετά θα είναι επικεφαλής της γραμματείας για την αγορά απασχόλησης. Πολύ λυπόμαστε γι' αυτό βέβαια, εις βάθος, γιατί είναι κρίμα να χάσουμε τη Σαμπίνα. Θα μας λείψει. Είναι ένας άνθρωπος στον οποίο μπορούσαμε πάντα να βασιστούμε, πάρα πολύ επαγγελματική αντιμετώπιση της και πραγματικά έχει τόσε πολλές γνώσεις για τον τρόπο εργασία του Κοινοβουλίου και εργάστηκε τόσο σκληρά για τη δική μα Επιτροπή. Συνέβαλε στην ανάπτυξη των μεθόδων εργασία τη επιτροπή. Έτσι μπόρεσε η Επιτροπή μας να αποκτήσει πραγματικά πάρα πολύ σημαντική θέση Μπορέσαμε να εξετάσουμε πολλά θέματα νομοθετικά και συμβάλαμε ούτω ώστε το gender mainstreaming να περάσει στην ημερησία διαδέκτου του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ λοιπόν για όσα κάνατε για την Επιτροπή μας και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην περαιτέρω σταδιοδρομία σας. Και θα μπορούσαμε, εάν χρειαστεί, να έχουμε πάρα πολύ καλές επαφές και συνεργασία με την Επιτροπή Απασχόλησης ε, στην περίπτωση αυτή. Ελπίζω πολύ από εσά σήμερα το βράδυ στις 6.30 να είναι παρόντες και παρούσες ε, σε αυτή τη μικρή δεξίωση για τον αποχαιρετισμό της Σαμπίνα που θα μπορέσουμε και κατηδία να την ευχαριστήσουμε για όσα έκανε για μας. Eh, eh, eh, Θα ήθελα τώρα να συνεχίσω με τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου και τις συστάσεις των συντονιστών. Πήρατε νομίζω ένα εγγραφό σχετικό. Περνάμε στο σημείο 7 τώρα. Equality between women and men in Europe, Union, okay. Ισότητα των γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Εντφέλντ. Yes, thank you, Chair. Uh, good morning. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ε, γνωρίζετε, 236 τροπολογίες έχουν κατατεθεί στην έκθεσή μου και όταν ξεπέρασα το αρχικό σοκ παρατήρησα ότι περισσότερες εξ αυτών είναι ιδιαίτερα επικοδομητικές τροπολογίες ε, πολύ υψηλός αριθμός τροπολογιών ασχολείται με ζητήματα απασχόλησης και οικονομικής φύσης. Έχω κυκλοφορήσει προτάσεις για 19 συμβαστικές τροπολογίες, οι οποίες ομαδοποιούν τις τροπολογίες που αφορούν στο ίδιο ζήτημα. Θα βρείτε αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες στο έγγραφό σα. Δεν είχα τη δυνατότητα να τη συζητήσω αναλυτικά με τους κοιόδης ηγητές και εισηγήτριες, αλλά φαντάζομαι θα το πράξω συντόμω Σε ό,τι αφορά τώρα τις αναπομείνωσε τροπολογίες, μπορώ να δεχτώ ένα πολύ μεγάλο αριθμό αλλά προφανώς υπάρχουν κάποια θέματα επί των οποίων υπάρχουν διστάμενες απόψεις και για τα οποία θα χρειαστεί να ψηφίσουμε οι τροπολογίες μπορούν να ομαδοποιηθούν γύρω από τα παρακάτω θέματα, όπως σας είπα, ε, ότι έχει σχέση με την απασχόληση, την οικονομική κρίση, τη στρατηγική 2020 κλπ. Ε, αυτά αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των τροπολογιών. Υπάρχουν επίσης τροπολογίες για την βία, την οικογενειακή βία, ε, την βία κατά των γυναικών, θέματα περίθαλψης, ε, άδειε μητρότητας, υπάρχουν που αφορούν στις γυναίκες στις θέσεις ε, οι οποίες ε, αφορούν στη λήψη αποφάσεων. διακρίσεις, πολλαπλές διακρίσεις στις ε, στην γύρανση, θέματα ε, αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας. Όπως σας είπα, μπορούμε να βρούμε κάποιες συμφωνίες επί των σημείων αυτών. Τα πιο επίμαχα θέματα αφορούν τα σεξουαλικά δικαιώματα και δικαιώματα αναπαραγωγής απευθυνόμενη στο τηλέφωνο της ε, Λέγης ε, η Μιλήτρια. Ε, επίσης ζητήματα που άπτονται των αδειών μητρότητας και εδώ υπάρχουν διστάμενες απόψεις και θα χρειαστεί να ψηφίσουμε και τέλος θέματα από των οποίων μπορούμε να συμφωνήσουμε και αφορούν στις παραγράφους για την βοήθεια κατοίκων Δεν ξέρω, ίσως ε, να μην έγινε απόλυτα κατανοητή, ε, μην γνωρίζουν όλοι το ζήτημα εξαντλητικά. Θα δούμε αυτά ως εισαγωγή. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Συγγνώμη, υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Δυστυχώς ε, το... Όχι, όχι, συνεχίστε να μιλάτε τη γλώσσα σας. Απλά υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα, παρατηρεί ο Πρόεδρος. Λοιπόν, να ξεκινήσω από την αρχή. Συγγνώμη που η έκθεση αυτή είναι τόσο σημαντική και αναλυτική αλλά και ουσιαστική για την Επιτροπή μας και για το Κοινοβούλιο αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έφτασε με καθυστέρηση στα χέρια μας δεν ε, φταίει η συγγήτρια και ε, η κατρική ημερομηνία κατάσταση τροπολογιών ε, ορίστηκε πολύ νωρίς, ε, σε μεταφράσει όμως τη λάβαμε με καθυστέρηση. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να αποφύγουμε από εδώ και στο εξή. Τώρα η έκθεση, όπως σα είπα, είναι αναλυτική. Η συγγήτρια επικεντρώνεται σε ζητήματα τα οποία θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικά, αλλά η ομάδα μου, στην οποία εγώ είμαι και σκιώδη συγγήτρια, θεωρούμε ότι έχει πολλές ελλείψεις. Δεν είναι ότι δεν μας αρέσει αλλά το γεγονός ότι υπάρχουν 236 τροπολογίες αυτό δείχνει ότι υπάρχουν ελλείψεις. Η συγγήτρια όμως ε, ελπίζουμε θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να βελτιώσει την έκθεσή της. Εμείς μπορούμε να δεχτούμε τις περισσότερες από 19 συμβασικές τροπολογίες και ελπίζω πως ε, θα τροποποιηθεί κατά το επιθυμητό η έκθεση και έτσι θα μπορέσουμε να την υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Ευρώπα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω για την εργασία σας ε, κυρία Ίνβελτ. Ε, περίπου 240 τροπολογίες ε, όπως είπατε υπάρχουν. Είδαμε ότι τα θέματα που μας, αφορούν, μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα είναι αυτά της απασχόλησης, η βία κατά των γυναικών, το ζήτημα της ε, εργασίας, ε, της παιδικής εργασίας. Η Επιτροπή μας θα πρέπει να ασχοληθεί με όλα αυτά τα ζητήματα και να τα προωθήσει, διότι πολλές κυβερνήσεις ε, δεν κατανοούν τι σημαίνει εργαζόμενη γυναίκα και παράλληλα μητέρα. Οι συμβαστικές τροπολογίες είναι κάτι με το οποίο μπορούμε από ό,τι φαίνεται να συμφωνήσουμε. Τα ζητήματα τα οποία θίξατε μας ενδιαφέρουν άμεσα και σας ευχαριστώ για την εργασία σας και θα τα πούμε στις συνεργίες των σκιωδών εισηγητών. Η κυρία Νέλη Σουέβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να χαιρετήσω το ε, δουλειά της εισηγήτριας. Δεν θα επαναλάβω τα όσα υπόθηκαν, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στις τροπολογίες που έχω καταθέσει. Βλέπω ότι έχουν συμπεριληφθεί συμβαστικές τροπολογίες. Ε, Παρατήρω και εγώ ότι τις λάβαμε με ιδιαίτερη καθυστέρηση και θα ήθελα να επανέλθω όμως πάνω σε έξι σημεία. Οι τροπολογίες μου αφορούσαν σε πολύ ε, συγκεκριμένα ζητήματα που κατά την μου έλειπαν από την έκθεση και σήμερα από το του σύμβασμό πιστεύω όλοι να συμφωνήσουμε. Όλοι συμφωνούμε επίση με τη συγκήτρια όταν δηλώνει ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στην πολιτική εκπροσώπηση των γυναικών και η τροπολογία με παρθμό 34 αφορά αυτό το σημείο. Διαπιστώνω ότι είναι αντικείμενο τροπολογία συμβαστική 11 και διαπιστώνω ότι σε πολλά κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόμαστε σε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, 15%. Είναι πολύ χαμηλό λοιπόν το ποσοστό αυτό. Δεύτερον, διαπιστώνω ότι έχει συμπεριληφθεί στην υπαριθμό 1 βασική τροπολογία, τροπολογία 42 και 151 οι ε, τροπολογίες ε, αυτές ε, αφορούν ζητήματα τα οποία δεν εξετάζει εκτενώς η έκθεσή της, αλλά είναι σημαντικά θέματα η οικονομική και ψυχολογική βία. Όταν μιλάμε για οικογενειακή βία, πολύ γρήγορα κάνουμε τη συσχετισμό με την φυσική βία. Η φυσική βία φυσικά είναι ουσιαστική, 20-25% των γυναικών υφίστανται οικογενειακή βία, αλλά δεν αφορά μόνο την οικογενειακή βία, αλλά ασκείται και ψυχολογική βία, ασκώντας πίεση στον ε, σύντροφο, να ε, σε οικονομικά ζητήματα, να μην ε, δίνει χρήματα κλπ. Αυτή η οικονομική βία λοιπόν είναι πολύ σημαντική και χαίρομαι που έχει συμπεριληφθεί στην συμβαστική τροπολογία. Τέλος, τα τρία τελευταία σημεία. Φυσικά η τα νηπιαγωγεία και η παιδική σταθμή είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Βλέπω ότι έχει συμπεριληφθεί στην συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 7 και στην υπαριθμών 5 συμβαστική τροπολογία υπάρχει το θέμα των οικονομία και των νέων τεχνολογιών και για να παραμείνουμε στους, στην εποχή μα. το ζήτημα θα πρέπει να το εξετάσουμε και να μην το παρακάμψουμε. τέλο κάτι το οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί στι συμβαστικέ τροπολογίε και θα ε, πρέπει να γίνει ε, αναφορά στην βία ως ε, όπλο ε, σε περίοδους πολέμου θα πρέπει λοιπόν να το εγγραφεί και στις προτεραιότητες διότι πρόκειται για ένα ζήτημα που αποτελεί μάστιγα σε διάφορες περιοχές του κόσμου και έτσι θα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα προς τις γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί βιασμού. Σας ευχαριστώ λοιπόν, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια για την ε, πολύ καλή και σε βάθος εργασία της. Ε, ευχαριστώ. Δεν βλέπω να επιθυμεί κάποιος άλλος να λάβει το λόγο. Είναι η συγγήτρια. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους ε, σε ό,τι φορά το ζήτημα το μεταφραστικό. Είναι ένα κλασικό θέμα. Συμβαίνει από καιρούς καιρών, ε, δεν είμαι υπεύθυνη κατανοώ ότι είναι δύσκολο να δουλέψει κανείς κάτω από αυτές τις ε, συνθήκες. Εντάχει λοιπόν να αναφερθώ στα σχόλια. της ομάδας ε, ε, S&D για τον χρόνο, για τον χώρο. Έχουμε μόνο τέσσερις σελίδες, δεν μπορούσαμε να τα συμπεριλάβουμε όλα. Τα στοιχεία λοιπόν των τροπολογιών, όπως σας είπα, στι περισσότερε περιπτώσει με βρίσκουν σύμφωνοι και θα φροντίσω να τα συμπεριλάβω. Τώρα η κυρία Ιρούκα ε, τόνισε κάποια ζητήματα, χωρίς όμως ε, να εγείρεζε ερωτήματα η κυρία Βερτσέβα. Ναι, συμφωνώ σχεδόν με όλα όσα είπατε, εκτός από ένα. Η ψυχολογική και οικονομική βία. Μόλον ότι αναγνωρίζω την σοβαρότητα των προβλημάτων που θίξατε. Ξέρω ότι είναι σοβαρό, αλλά δεν θα τα συνδέσω με το ζήτημα της βίας, διότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έναν, κάποιες πληθωριστικές τάσεις σε ό,τι φορά την χρήση του όρου βία. Τώρα για το τελευταίο σας σημείο για τη βία ως ε, εργαλείο πολέμου. Το άφησα εκτός ε, των συμβαστικών τροπολογιών, ε, αλλά θα ζητήσω να υπερψηφιστεί. Συμφωνώ μαζί σας, η Γραμματεία ετοιμάζει έναν κατάλογο ψηφοφοριών και θα τον μοιράσουμε το συντομότερο. Ελπίζω να λάβω τις αποφάσεις των συντακτών τροπολογιών ε, περί του καταλόγου. Δεν μπορώ φυσικά να συμπεριλάβω όλες τις τροπολογίες και όλα τα ζητήματα που εθίγησαν. 85 τροπολογίες ε, κάλυψα με 19 συμβαστικές τροπολογίες και Ίσως ε, να υπάρχει χώρος ε, για κάποιες περαιτέρω συμβαστικές τροπολογίες ε. Λοιπόν, πολλά ζητήματα γέρθησαν και θα κυκλοφορήσω, κυκλοφορήσω την κατάλογο των ψηφοφοριών το συντομότερο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επισημάνω ότι θα ψηφίσουμε από αυτή τη ε, γνωμοδότηση 27 και 28 Ιανουαρίου, ε, Φεβρουαρίου συγγνώμη, και θα περάσει την Ολομέλεια τον Απρίλιο. Περνάμε στο σημείο 8. γυναίκες και εγκληματική αλλαγή. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Κινλίσεν, εισηγητρία. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Εφόσον αυτή τη στιγμή είμαστε σε προηγούμενο στάδιο σχέση με την ε, συνάδελφο. Έχουμε λάβει περίπου 50 τροπολογίες που είναι πολύ θετικέ και εμπλουτίζουν ε, την έκθεση, ε, η οποία τη χάνει συνένεση από ό,τι καταλαβαίνω. Θα ήταν καλό τώρα να θέσουμε μια ημερομηνία για να συνεδριάσουν οι σκιώδεις, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα. Δεν ήθελα να πω κάτι πιο συγκεκριμένο, θα ήθελα να ε, να συναντήσω τους ανθρώπους που έχουν υποβάλει τις τροπολογίες αυτές, να συναντηθούμε λοιπόν και να καταλήξουμε σε συμβασμούς που σίγουρα θα είναι εύκολο να βρεθούν. Ευχαριστώ και πάλι όμως τους συναδέλφους ε, για την εμπλουτιστική του δράση. Ευχαριστώ κυρία Στρέλα. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Συμφωνώ με την εισηγητρία. Θα ήταν καλό να συναντηθούμε και να καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικέ προτάσεις. Και εγώ υπέβαλα ορισμένες ε, τροπολογίες εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας των σοσιαλιστών. και είμαι διατεθειμένη να συνεργαστώ μαζί σας και με τους άλλους αισκαιώδεις εισηγητές από τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες. Ούτως ώστε να επιτύχουμε συνένεση και να μεριμνήσουμε ώστε η έκθεση αυτή να μας εκπροσωπεί όλους. Δεν θα μιλήσω πιο συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή για τις τροπολογίες μου, αφόσον θα τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστώ. Ε, από ό,τι βλέπω δεν θέλει κάποιος άλλος το βήμα. Εγώ ως εσκιώδης Θα ήθελα να πω και εγώ ότι πρόκειται για εξαιρετική έκθεση. Καλύπτει πολλά σημεία και οι τροπολογίες δείχνουν, όπως είπατε, ότι συμφωνούμε και ότι λογικά δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Θα είναι μάλλον εύκολο να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Συμφωνώ λοιπόν με την ε, πρότασή σας να κάνουμε μια συνεδρίαση για να τα συζητήσουμε. Και αυτή η έκθεση θα είναι ιδιαίτερα καλή και θα καλύπτει πολλά σημαντικά ζητήματα. Και χαίρομαι που ε, καλύπτει τόσο ευρύ φάσμα τομέων ε, σε ό,τι φορά την διασύνδεση ε, της κλιματικής αλλαγής και της διάστασης του φύλου. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Κανείς άλλος δεν θέλει να πάρει το λόγο. Τέλος λοιπόν για το κλείσιμο κυρία Κιλνίσεν. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Χαίρομαι ιδιαίτερα ε, που υπάρχει τόσο θετική στάση ε, για ένα ζήτημα που βεβαίως είναι θεμελιώδης σημασίας και είναι δύσκολο να περάσει στην κοινή γνώμη ευρύτερα. Όταν μιλάμε για την ε, κλιματική αλλαγή και τη φυλετική διάσταση, πάντα αυτό είναι κάτι που αντιμετωπίζει δυσκολίες, οπότε σας ευχαριστώ για τη στάση σας. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Όπως ξέρετε, στην Επιτροπή η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών ήταν η 10η Ιανουαρίου. Εμείς θα συζητάμε εδώ σήμερα και η Επιτροπή θα ψηφίσει από αυτόν στις 27-28 Φεβρουαρίου και στην Ολομέλεια θα περάσει είτε τον Μάρτιο είτε τον Απρίλιο. Φτάνουμε λοιπόν τώρα εφόσον πάμε τόσο γρήγορα δεν ξέρω πώς να το τραβήξω δεν ξέρω τι να κάνω ακριβώς αυτή τη στιγμή αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ώρα της συνεδρίας των συντονιστών Καλό θα ήταν λοιπόν να σταματήσουμε εδώ και να ξεκινήσουμε και πάλι στις 3 το απόγευμα όταν θα έρθουν οι Υπουργοί ε, της Δανικής Προεδρίας. Στις 3 λοιπόν και στις 11 και 4 η συνεδρία των συντονιστών. Θέλω να είστε πολύ ακριβείς ε, γιατί πρέπει να συζητήσουμε πολλά σε αυτή τη συνεδρίαση. Σταματούμε εδώ λοιπόν. Οι συντονιστές στις 11 και 4 και οι υπόλοιποι στις 3.